Εδώ, εδώ στην πρώτη σειρά είναι για σας κρατημένη. Ich eröffne die Sitzung, die eine außerordentliche Sitzung. Κυρίσω την έναρξη της έκτακτης συνεδρίας της Επιτροπής μας. Maria hatte den Η Μαρία είχε κάνει την πρόταση το σημείο 7 να το αλλάξουμε το 8, αλλά εμείς θα προτιμούσαμε να τηρήσουμε τη σειρά μας. Ε, θα προλάβουμε. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε τελειώσει και διεκπαιρώσει τα θέματα μέχρι τις 6.30 αν δουλέψουμε σωστά. Σας επισημαίνω το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα εδώ να έχουμε web stream. Δηλαδή, όλοι εκείνοι που θεωρούν ότι όλα αυτά που λέμε θα πρέπει να ανατιστούν για τον αιώνα τον άπαντα, θα βγει στο web stream, στο διαδίκτυο δηλαδή, και αυτό δείχνει πόσο ε, ε, δεδομένη είναι η διαφάνεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, για την ημερήσια διάταξη έχετε άλλες επιθυμίες. Όχι, από ό,τι βλέπω. Και μπορούμε να θεωρήσουμε το σημείο 3, κοινωνική ευθύνη. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Ε, η συγκεκριτή είναι ο κύριος ε, Θα πάρει το λόγο όμως ένας συνάδελφος από τις κάτω χώρες διότι απουσιάζει ο εισηγητής. Έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Τόμας. Θα πω λίγα λογάκια για την έκθεση Λιτίνεν. Η έκθεση βεβαίως αυτή δεν είναι μεμονωμένη, υπάρχει σαφή σχέση με μεταξύ άλλων την έκθεση που συζητάμε αυτή τη στιγμή και αφορά την καταπολέμηση της ε, παρανομίας και έχουμε αρκετές ε, ήδη εκθέσεις για αυτό το, το θέμα που έχει συζητήσει το Κοινοβούλιο. Το πρόβλημα εδώ πέρα που μας απασχολεί είναι ότι έχουμε την αύξηση των ε, υπεργολάβων και την λεγόμενη εξωτερήκευση, το outsourcing συγκεκριμένων λειτουργιών της αλυσίδας παραγωγής. Το ζήτημα λοιπόν όχι μόνο της εταιρική κοινωνικής ευθύνης, αλλά και το ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνος, ο συνομιλητής, αν θέλετε, στον κοινωνικό ε, τομέα. Ένα θέμα που γίνεται όλο και πιο οξυμένο και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πως ε, οι λύσεις τις οποίες εξετάζουμε πηγαίνουν σε δύο κατευθύνσεις. Η μελέτη του συναδέλφου Λετίνε αναφέρεται στις εμπειρίες ε, που, 8 ε, χωρών στον τομέα της οικοδομής. Μιλάει αφενός για την ε, αλυσίδα, ένα θέμα το οποίο είναι εδώ και χρόνια σημαντικό. Μια άλλη λύση η οποία έχει επιλεχθεί και αναφέρεται είναι ο λεγόμενος κώδικας συμπεριφοράς και το τι περιέχεται εκεί πέρα. Το οποίο αφορά παραδείγματος χάρη τους εργαζομένους ε, πολιεθνικών και μεταξύ άλλων εκεί πέρα αναφέρεται πως οι εργαζόμενοι έχουν ε, εγγύηση για όλες τις, ε, τα κοινωνικά τους δικαιώματα του που δραστηριοποιείται και αυτό δεν ε, περιορίζεται μόνο στον τομέα της οικοδομής αλλά και σε εταιρείε που παρέχουν υπηρεσίες κοινή ωφέλεια, όπως παραδείγματο χάρη των, των υδάτων και αυτό γίνεται μέσω της κατανομής δραστηριοτήτων σε υπεργολάβους ή σε προμηθευτές. Το δύσκολο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει εδώ πέρα ο συνάδελφος είναι η καινοτομία την οποία πρέπει να εισαγάγουμε στην νομοθεσία και συμφωνώ με το συμπέρασμά του πως ε, η κοινωνική ευθύνη υπάρχει και πρέπει να ρυθμιστεί εκεί πέρα όπου έχουμε μία λυσίδα παραγωγής και έχουμε ένα πακέτο ολόκληρο ε, τροπολογιών οι δε συζητήσεις ε, γίνονται σχετική επιτροπή, όπου δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε εδώ πέρα. Ε, τα πράγματα είναι νομίζω και τα σημάδια προφανή κατά την απόψη μου. Now we have time for discussion. Λοιπόν, τώρα έχουμε χρόνο συζήτησης. Steven Hughes. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να αφαιρθώ σε άλλη μια πτυχή της έκθεσης αυτής. Ε, ο κύριος Λέτνεν ζητά συγγνώμη. Ε, είναι απόν, γι' αυτό τον εκπροσώψει ο Γιάν. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ασχολείται με την έκθεση ΦΑΒΑ για την παράνομη εργασία που ανέφερε ο Γιάν και υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί προτείνουν να υιοθετήσουν μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση που συμπεριλαμβάνει η τροπολογία στο άρθρο 9 που θα περιορίσει την αστική ευθύνη μόνο στο πρώτο στρώμα, εάν θέλετε, υπεργολαβίας. Οπότε ε, θα χειροτερέψουν τα πράγματα αντί να καλυτερεύσουν και είναι σαφής η ανάγκη για αυτή την έκθεση. Η Λίμπε πιέζει πάρα πολύ για να πάει αυτό στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα, κάτι το οποίο θα υπονομεύσει αυτή την έκθεση πριν πάει καν στην Ολομέλεια. Ίσως η γραμματεία μπορεί να έρθει σε επαφή με τη γραμματεία της Λίμπε για να δει εάν ε, μπορούμε να αναβάλουμε την άλλη έκθεση για να ξεκαθαρίσει αυτό το χάλι. Δεν υπάρχει λόγο για να συμφωνήσουμε από τώρα, από την πρώτη ανάγνωση. Είναι σοβαρό το ζήτημα και πρέπει να το δούμε την ισχύα μα. Äh, να το δουν αυτά οι πρόεδροι μεταξύ τους, γιατί αν κάνουμε τη δουλειά δεν θα πρέπει να είναι μάταιοι δεν μπορούμε να είμαστε εκπρόθεσμοι. 66 τροπολογίες έχουμε καταθέσει εμεί που θέλουμε να συζητήσουμε εύστοχα έτσι και είχαμε προγραμματίσει η έγκριση είναι στις 11 Φεβρουαρίου και μετά στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Ας το δουν αυτό παρακαλώ οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους να, να κερδίσουμε λίγο χρόνο αν γίνεται. Γιατί είναι κρίμα να κάνει δουλειά μια ε, επιτροπή και να μην λαμβάνεται υπόψη αυτή η δουλειά. Είναι, είναι και ο χειρότερο δρόμο. Καλά, είναι και έκθεση πρωτοβουλία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μερικοί θεωρούν ότι οι εκθέσεις πρωτοβουλία είναι τελείω άχρηστε και χωρί συζήτηση θα πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία επιτέλου κάποια στιγμή και βοηθήστε. Γιατί είναι πραγματικά γελίο. Πρέπει να συζητάμε. Πρέπει να συζητάμε επί το περιεχομένου. Χωρί συζήτηση δεν το κάνουμε. Παραμένει μόνο κλειστός κύκλος των επιτροπών. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Σχόλια. Ε, είχε κάνει ο κύριος Λέχτινεν για τις τροπολογίες Γιάννη, σου είχε πει τίποτα. Όχι. Καλά. Ας φροντίσουμε λοιπόν να ξανασυζητήσουν οι δύο πρόεδροι των επιτροπών. Ε, εντάξει, συμφωνούν όλοι και πάμε στο επόμενο θέμα. Sind ε, die Έχουμε τα θέματα, τα δικαιώματα των ασθενών, μια νομοθετική έκθεση, δηλαδή πολύ σημαντική έκθεση του συναδέλφου Μπραγκέτο, που έχει τη δυνατότητα να μας ε, αναφέρει εδώ πέρα. Σχετικά έχουμε 184 ε, τροπολογίες και νομίζω ότι μπορεί να γίνει πολύ συναρπαστική αυτή η υπόθεση. Έχουμε συνολικά 206. Ε, τι, τι ωραία πράγματα έχει κάνει εκεί πέρα και ενδιαφέρει τους πάντες τόσο πολύ αυτή η έκθεση. Έχεις τον λόγο. Ο Αυτό δείχνει την τεράστια σημασία που έχει αυτή η έκθεση. Όχι τόσο για τη δική μας Επιτροπή, για την καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή. Αλλά η συζήτηση που έγινε με αφορμή αυτής της νομοθετικής πρότασης είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και σε αυτή την Επιτροπή έγινε επίσης μια συζήτηση με θετικό πνεύμα και οι 200 τροπολογίες επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτή τη σημασία της έκθεσης. Δεν θα σας απαριθμίσω τις τροπολογίες αλίμονο, τις έχω ομαδοποιήσει σε βασικές κατηγορίες. Κάποιες τροπολογίες ε, θέλουν απλώς να διευκρινίσουν αφιλεγόμενα σημεία ή σημεία που επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες. Κάποιες άλλες τροπολογίες θέλουν να τονίσουν τις ανησυχίες για τις εγγύησεις που πρέπει να προσφέρουμε στους ασθενείς. Αυτές οι τροπολογίες με τους κατάλληλους συμβιβασμούς μπορούν να γίνουν δεκτές στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Υπάρχουν βέβαια κάποιες άλλες τροπολογίες που θέλουν να μειώσουν το πεδίο εφαρμογής, την εμβέλεια της οδηγίας. Και προφανώς αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Συνοπτικά λοιπόν να σας πω ότι η πρόταση γίνεται θετική, γίνεται, τη, δεχόμαστε με ευνοϊκό πνεύμα, πέρα από την απόφαση του 10. Δεύτερον, πολλές τροπολογίες υπενθυμίζουν τον ουσιαστικό ρόλο των υγειονομικών υπηρεσιών στο κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο και υπενθυμίζουν και την ε, ανάγκη να υπάρχει προσπελασιμότητα των υπηρεσιών αυτών, καθολικότητα, ποιότητα, ισότητα, αλληλεγγύη. Επίσης υπενθυμίζουμε την ε, ασφάλεια των εργαζομένων Ξεκίνησε μάλιστα μια συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Επιτροπή για το θέμα των νοσοκομιακών λοιμόξεων και κάποιες τροπολογίες ακριβώς αντανακλούν αυτές τις ανησυχίες που μου φαίνονται πολύ σωστές. Όπως επίσης μιλάνε για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση ε, μεταξύ της συνεργασίας ε, συνεργασία των περιφερειών. Γιατί σε πολλά κράτη-μέλη την αρμοδιότητα την έχουν περισσότερο οι περιφέρειες και όχι τόσο τα κράτη. Επομένως, ο διασυνοριακός χαρακτήρας και η συνεργασία μεταξύ των περιφερειών είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ένα αρκετά αμφιλεγόμενο σημείο, το οποίο όμως πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε, για το οποίο να μπορούμε να βρούμε λύση, είναι η προληπτική έγκριση από πλευρά κρατών μελών. Που να είναι όμω ευέλικτη προ όφελο του ασθενού. Και παράλληλα να δώσει και τη δυνατότητα στους υπεύθυνους για την υγειονομική διαχείριση και το προγραμματισμό των υπηρεσιών σε νοσοκομιακό επίπεδο να οργανωθούν όπως θέλουν. Κάποιες τροπολογίες μιλάνε για την ενδυνάμωση του στοιχείου της πληροφόρησης και αυτό επίσης ε, νομίζω ότι είναι αποφασιστικό στοιχείο. Μπορούν οι πολίτες να υποφεληθούν από αυτή την πληροφόρηση. Υπάρχουν τώρα κάποιες τροπολογίες που θέλω να ενσωματώσω και που μιλούν για την ανάγκη ε, σύνδεσης με το κανονισμό ε, για τα κοινωνικά καθεστώτα, κοινωνικά συστήματα μάλλον, ορισμένες τροπολογίες μιλούν για διευκρίνηση των ορισμών. Όπως παραδείγματο χάρη τι είναι η υγειονομική περίθαλψη και τι είναι η νοσοκομιακή περίθαλψη. Προσοχή σε αυτό το σημείο δεδομένης και της αρμοδιότητας της ε, Επιτροπής μας, η οποία δεν είναι εκεί πλέον αρμόδια. Δεν μπορούμε να μπούμε εμείς ε, στην ουσία των ορισμών, που είναι υγειονομικού χαρακτήρα. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές ομαδοποιημένες πάντα οι τροπολογίες που έχουν μεγαλύτερη σημασία και επί των οποίων μπορούμε να εργαστούμε, ούτω ώστε να βρούμε αποδεκτούς συμβιβασμούς, προκειμένου αυτές οι 200 τροπολογίες να ενταχθούν όσο γίνεται στην πρόταση. Η πρόταση βέβαια πρέπει να παραμείνει και ευέλικτη και σωστή έτσι από γλωσσική άποψη. Δεν μπορούμε να τη βαρύνουμε πολύ τη διατύπωση της πρότασης. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής βλέπω θέλει να δεχτεί αρκετές τροπολογίες εκτός από μερικές. Μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα. Η Λίζ είναι η σκιώδης εισηγήτρια για τους φιλελεύθερους. Λίζ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για τη δουλειά που έχετε κάνει σε αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε έχω καταθέσει μια σειρά τροπολογιών και σας ευχαριστώ που λέτε ότι σε γενικές γραμμές συμφωνείτε με τις περισσότερες. Απλά να τις διατρέξουμε η 39 κάτι το οποίο απασχολεί εμένα και τον Στίβεν Χιούς. Μια τροπολογία για τους ε, τραυματισμούς από βελόνες και σύριγγες όσον αφορά τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Ε, θα ήθελα να αναφέρετε κάτι σχετικό για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις ε, όπως την τροπολογία 4087. Πρέπει να διασφαλίσουμε κάθε, ότι κάθε εργαζόμενο στον τομέα της υγείας σε κάθε κράτος μέλος είναι ικανός. Και πρέπει να υπάρχει διαβεβαίωση στους ασθενείς πως ε, οι εργαζόμενοι στην τομέα της υγείας έχουν ένα ίδιο βαθμό επαγγελματικής επάρκειας σε κάθε κράτος μέλος. Επίσης, για την 168, 179 και 190 να υπάρχει ένας μηχανισμός αποζημίωσης και κάποιο είδος προσφυγής εάν πηγαίνουν τα πράγματα στραβά. Δηλαδή αν χάσουν ε, την ε, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ε, κάποιοι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας σε ένα κράτος μέλος να το ξέρουν και στα άλλα κράτη-μέλη για να μην τους απασχολούν 5472 για την πρόσβαση από τους αναπήρους και για την 101. Μιλάτε για τις συνταγές. Ξέρω πως κάποια κράτη-μέλη έχουν συνταγές ε, ειδικέ για ανάπηρους ε, με την έννοια ότι μπορούν να δουν αυτές τις προφορίες και χρησιμοποιείται να έχουμε και κάτι εδώ πέρα. Επίσης για την προκαταβολή των εξόδων ε, και την πρώτερη εξουσιοδότηση. Αυτό μάλλον θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στο 154 όπως ξέρετε προσπάθησα να βρω μία μέση οδό μεταξύ κάποιων τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Δηλαδή αυτή η πρώτη εξοδότηση μπορεί να δοθεί στους ασθενείς και το... τα μετρητά να δοθούν, να προκαταβληθούν από το κράτος μέλος εάν θα ήταν η ίδια θεραπεία και το ίδιο κόστος και στο κράτος μέλος τους, δηλαδή να είναι οι ίδιες οι υπηρεσίες. Δηλαδή, όπως λέμε εδώ πέρα, ότι θα μπορούσαν να πληρωθούν με τον ίδιο τρόπο εάν αυτό γίνονταν στο σύστημα υγείας του κράτους μέλους τους. Και άρα μπορεί τα χρήματα να μεταφερθούν απευθείας από το κράτος μέλος. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την ε, δουλειά σας. Αυτά ήταν τα πιο δύσκολα σημεία και γνωρίζω πως συνεργάζεστε και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και εγώ εντός της ομάδας μου και θα έχουμε μια πολύ καλή έκθεση, αλλά υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα που πρέπει να γίνει για να χτενίσουμε κάποια πράγματα και αυτή η πρώτη εξοδότηση είναι ένας από τους βασικούς τομείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, όλες. Άννα Φελάνγκρα μετά έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το ότι υποσχέθηκε πως θα συνεργαστεί με τους κοιόδης εισηγητές ε, και νομίζω πως ε, θα έχουμε αρκετά καλές ε, ε, τροπολογίες. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μας, αλλά όταν κοιτάω τις τροπολογίες νομίζω ότι πρέπει να καθυσυχαστούμε σε κάποια σημεία. Υπάρχουν πέντε κρίσιμα ουσιαστικά πολιτικά σημεία που θέλω εγώ να αναφέρω. δεν ξέρω εάν η Επιτροπή μας, η Γραμματεία μας έχει έρθει σε επαφή με την κύρια Επιτροπή εδώ πέρα, την Επιτροπή Περιβάλλοντος δηλαδή. Και το ρωτάω για το εξής. Εγώ παρατήρησα και θα το παρατήρησε και ο εισηγητής πως πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν εργαστεί στα άρθρα μετά τα άρθρα 10 και 11. Δηλαδή αυτά τα οποία αφορούν το e-health, συνεργασία κρατών μελών, στον τομέα της παροχής υγείας. Έχουμε εδώ πέρα ένα ζήτημα κλειδί που πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν ψηφίσουμε που σταματάει η αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Δηλαδή αν το δούμε στενά, εγώ αντιλαμβάνομαι την κατάσταση ως εξής. Εμείς φτάνουμε μέχρι το σημείο του να υπάρξει κάποιος συντονισμός και όχι να δούμε ποια είναι η ποιότητα της παροχής υγείας. Δεν είναι δική μας ε, αρμοδιότητα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του κυρίου Μπόβης νομίζω. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε πού στέκεται ακριβώς η Επιτροπή μας και να ενισχυθούμε λίγο κάπως όσον αφορά τις αρμοδιότητές μας. Και τώρα κάποια άλλα ζητήματα, κλειδιά που πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Το πρώτο αφορά τη νομική βάση αυτής της οδηγίας. Έχω καταθέσει μια σειρά τροπολογίες και κάποιοι συνάλφοι Steven Hughes, Jan ε, Kremers ε, έχουν ε, πει πως πρέπει να βασιστούμε στο άρθρο 153, αυτό της συνθήκης δηλαδή που αφορά τη δημόσια υγεία. Βεβαίως, εάν το δούμε στενά, η Ευρώπη έχει μόνο έναν υποστηρικτικό ρόλο στον τομέα της δημόσιας υγείας, κυρίως για μεταδοτικές ασθένειες και τα λοιπά λοιμώδης, αλλά δεν θα είναι και άσχημο νομίζω να υπαχθούμε στο άρθρο 153 γιατί απομακρυνόμαστε από την καθαρή βάση της ελευθερίας, ε, της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ε, εσωτερικής ε, αγοράς. Και πηγαίνουμε πιο πολύ προς τα εκεί που θα θέλαμε να κινείται αυτό το κοινοβούλιο. Το ίδιο ισχύει και για την προσθήκη του άρθρου 16, δηλαδή προσθήκης γενικής οικονομικής σημασίας. Κοιτάξτε, αν το δούμε και αυτό στενά, δεν προσθέτει κάτι το ουσιαστικό στην πρόταση, γιατί το άρθρο 16, έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, αποτελεί τη νομική βάση δράσης κοινότητας. Αλλά μιλάμε πάλι για το πώς θα ξεκαθαρίσουμε καλύτερα τη φιλοσοφία μας ότι η δημόσια υγεία είναι μια υπηρεσία γενικού δημόσιου συμφέροντος που πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο παιδοποιότητας για όλους τους ε, πολίτες κοινότητας. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το εύρος αυτής της οδηγίας. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να έχουμε πάντα κατά νου πως ε, αυτή η οδηγία και να με συγχωρήσετε για αυτό που θα πω, να κοιτάξουμε πάρα πολύ ε, καλά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο, γιατί έχω την εντύπωση πως αυτό το οποίο κάνει το Συμβούλιο ε, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτά τα οποία σκέφτεται η Κομισιόν και νομίζω και οι πράσινοι και το Συμβούλιο παρατηρούν πως ε, εδώ πέρα δεν μιλάμε για επέκταση αν θέλετε διεθνή της ε, παροχής ε, υγείας αλλά αφορά την κινητικότητα ασθενών δηλαδή ο ασθενής να πάει σε ένα άλλο κράτος μέλος για να μπορέσει εκεί να απολαύσει υπηρεσίες υγείας και όχι τη μετακίνηση επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. Αυτό σημαίνει πως ε, βεβαίως το εύρος αναφέρεται στο άρθρο 1, αλλά πρέπει να δούμε κάποιους ορισμούς διαφορετικά. Οπότε σημαντικό είναι να δούμε πως ε, κάποιοι συναδελφοί, όπως ακριβώς και το Συμβούλιο, πρέπει να ξεκαθαρίσουν πως μιλάμε για την κινητικότητα ασθενών και τη διασυνοριακή περίθαλψη. Δηλαδή κινητικότητα ασθενών και τίποτα άλλο. Νομίζω κάλυψα το σημείο 2. Ένα τρίτο σημαντικό θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας και ίσως ελπίζω αύριο που θα συζητήσουμε τις συμβαστικές λύσεις είναι το τι θα γίνει με τον, με τον κανονισμό για τον συντονισμό. Δηλαδή νομίζω ότι θα επιβεβαιώσετε ότι και εγώ και το Συμβούλιο ή οι πράσινοι ή και άλλοι συνάδελφοι πρέπει να ασκήσουν πίεση έτσι ώστε αυτή η οδηγία να μην ε, καταργήσει τον ε, κανονισμό για τον συντονισμό, αλλά πρέπει να υπάρξει απλά μια προσαρμογή του εκεί που έχουμε τις ανάλογες ε, προτεραιότητες. Δηλαδή, ο κανονισμός βεβαίως δίνει πολύ μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα στους ασθενείς από τη μια οδηγία. Δεύτερον, ο κανονισμός δεν κάνει λόγο για προκαταβολές αλλά υπάρχει κάποιος μηχανισμός ε, αποζημίωσης και βέβαια ο κανονισμός είναι πολύ σαφέστερος από την οδηγία. όσον αφορά την ε, οργάνωση και χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας. Οπότε πρέπει στο προσκήνιο να βρίσκεται ο κανονισμός του συντονισμού και η οδηγία θα καλύπτει τις υπόλοιπες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον ε, κανονισμό. Πρέπει βεβαίως να είμαστε και συνεκτικοί και να υπάρχει η εγγύηση στους ορισμούς ότι μιλάμε για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτό είναι το μήνυμα του Συμβουλίου και αρκετών συναδέλφων εδώ πέρα στις ε, τροπολογίες, δηλαδή ότι ο ορισμός που υπάρχει στον κανονισμό είναι ευρύτερος από την πρόταση της ε, Κομισιόν και πρέπει να είναι ξεκάθαρο νομίζω το σύστημα έτσι ώστε να είναι λίγο πολύ ίδιος ο ορισμός εδώ πέρα με τον ε, κανονισμό για τον συντονισμό. Επίσης θα θυμούνται οι συνάδελφοι πως ε, η Κομισιόν αναφέρεται συγκεκριμένα στις υπηρεσίες που παρέχονται από τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και καλύπτονται από την οδηγία, την οδηγία του 2005. Πολύ περιορισμένος ο ορισμός και υπάρχουν εκτός από αυτά πάρα πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που είναι αναγνωρισμένοι νομικά στα κράτη-μέλη και μπορούν βεβαίως και με βάση τον κανονισμό να πληρωθούν αλλά δεν καλύπτονται εδώ πέρα. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να έχουμε έναν όσο δυνατόν πιο ξεκάθαρο ορισμό για το τι σημαίνει παροχή υπηρεσιών υγείας σε αυτή την οδηγία. Όσον αφορά τώρα την πρώτερη εξοδότηση θεωρώ πως καλό και ευχάριστο είναι που βλέπουμε ότι όλοι σε αυτή την Επιτροπή και στο Συμβούλιο ξεκαθαρίζουν πως τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν την δυνατότητα όταν μιλάμε για νοσοκομεία και για εξειδικευμένη ε, περίθαλψη να μπορούν να ορίζουν μόνο τους ποια είναι αυτή η περίθαλψη και να λένε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται πρώτερη εξιοδότηση. Το βλέπω αυτό στις ε, τροπολογίες των Πρασίνων, του συναδέλφου Μπραγκέτο, του συναδέλφου Κοχ και της κυρίας Παναγιωτοπούλου, Ντεζίρ, τις δικές μου και θα έλεγα και το Συμβούλιο έχει την ίδια άποψη γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όταν μιλάμε για νοσοκομεία και τέτοια παροχή υγείας είναι τόσο ευαίσθητα, τόσο ακριβά που πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τα κράτη-μέλη αυτό το εργαλείο για να ορίσουν τι είναι αφενός και δεύτερον να ζητήσουν αυτή την πρώτερη εξοδότηση. Επίσης, αντί για τη διαδικασία της επιτροπολογίας που προτείνει η Κομισιόν, η Κομισιόν προτείνει δηλαδή να στηθεί μια επιτροπή για να καταλήξει στον ορισμό της νοσοκομιακής περίθαλψης κτλ. με βάση τις ε, λίστες των κρατών μελών. Εγώ λέω να τα αφήσουμε όλα αυτά κατά μέρος, να μην πάμε καν στην επιτροπολογία εγώ θα έλεγα αντί να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα συστήματα των διαφόρων κρατών μελών, θα είναι ενδιαφέρον να κοινοποιηθούν οι κατάλογοι στην Κομισιόν, αλλά μην τις δώσουμε εντολή να προχωρήσει σε εναρμόνιση. Απλά να έχει αυτές τις πληροφορίες. Ένα άλλο σημείο που ήθελα να αναφέρω είναι κάτι το οποίο ανέφερε η κυρία Λίν και ο εισηγητής μας, δηλαδή το θέμα ποιος πληρώνει και πόσο πληρώνει. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ πως αυτό είναι το δυσκολότερο σημείο όλων όσον αφορά αυτή την οδηγία. Δεν βλέπω, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι πώς το πλαίσιο αυτής της οδηγίας όταν μιλάμε για κινητικότητα ασθενών που βασίζεται στα άρθρα της συνθήκης, μιλάνε για ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών κτλ πώς μπορούμε να φτιάξουμε και να συνδέσουμε εδώ πέρα ένα συνδυασμό ε, αποζημίωσης που υπάρχει στο πλαίσιο του κανονισμού. Κάνουμε μια καλή προσπάθεια μέσω των προκαταβολών να ορίσουμε ποιο είναι το επίπεδο από το οποίο καλύπτεται από το κράτος μέλος του ο ασθενής. Ε, είδα επίσης πως ε, η συνάδελφος Κρέτου μιλάει στις τροπολογίες της για ένα σύστημα καταβολής αποζημίωσης ε, μεταξύ των δύο κρατών μελών. Βλέπω επίσης πως ο Σνάλφος Μπόβη στην κύρια επιτροπή προτείνει να εργαστούμε με το σύστημα των κουπονιών, όπου υπάρχει βεβαίω πρώτερη εξουσιοδότηση και καλεί την Κομισιόν να βρει ένα τέτοιο μηχανισμό αντιστάθμισης. Για, για να αλήθεια, δεν θα λειτουργήσουν όλα αυτά γιατί αυτός εδώ πέρα δεν είναι ο κανονισμός του συντονισμού. Πώς δηλαδή θα λάβουν τα χρήματά τους ε, και τα έξοδά τους αυτοί οι οποίοι παρέχουν τις ε, υπηρεσίες τους όταν ε, λέει ο ότι εγώ αυτά έχω να πληρώσω. Βέβαια στην Ολλανδία υπάρχει ένα σχετικός μηχανισμός αλλά όταν μιλάμε για ένα μηχανισμό μεταξύ χωρών ε, πρέπει να σκεφτείτε ότι ορισμένα πράγματα καλύπτονται σε κάποιες χώρες, ορισμένα όχι άλλα. Και δεν ξέρω πώς θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα και είναι το μεγάλο πρόβλημα γιατί εδώ είναι η ουσία αυτής της οδηγίας. Η οδηγία αυτή μπορεί ε, και πρέπει να δώσει περισσότερη νομική βεβαιότητα σε ασθενείς που πάνε στο εξωτερικό για κάποια περίθαλψη αλλά δεν θα οδηγήσει ποτέ σε εξομοίωση αυτών των συστημάτων για τον απλό λόγο ότι σε κάποια, άλλα κράτη, σε κάποια κράτη-μέλη πληρώνει εκ των προτέρων, ο ασθενής σε κάποια άλλη όχι. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το, το ζήτημα. Εντάξει, έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες, αλλά η συζήτηση είναι ανοιχτή. Και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η προβληματική αυτή του inflow και του outflow, εισρωών και εκρώων θεωρώ πως η Κομισιόν και οι τροπολογίες εδώ πέρα έχουν δει πάρα πολύ καλά το σύστημα αυτών των εκροών που θα προκύψουν από τα συστήματα. Νομίζω πως οι τροπολογίες των πρασίνων το καλύπτουν το θέμα. Δηλαδή λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει πρώτερη εξουσιοδότηση και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που θα παίζει το ρόλο ενός ε, φύλακα αν θέλετε. Τώρα για τις εισρωές ε, δεν νομίζω να, είναι κάποιο, να υπάρχει κάποιος που έχει σκεφτεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά βεβαίως ε, εγώ προέρχομαι από μια χώρα η οποία αν θέλετε σε καθαρό αριθμό δέχεται περισσότερους ασθενές από τους στέλνει. Οπότε δεν έχει πρόβλημα. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει εάν γίνει πιο σίγουρη η κινητικότητα των ασθενών και θα υπάρχει μεγαλύτερη χρήση της. Οπότε έχω και αυτό το ερώτημα στον εισηγητή μας να δει τις τροπολογίες που έχω καταθέσει όσον αφορά τις ε, και το τι θα πρέπει να είναι τα μέτρα που θα λάβουν τα κράτη-μέλη. Αυτά νομίζω συνάδελφοι ήταν τα κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας στην άτυπη εργασία που θα ακολουθήσει και θα ήθελα Σα παρακαλώ πάρα πολύ η γραμματεία και εσείς να δείτε το ζήτημα των ομοδιοτήτων τη Επιτροπής μας για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, σε ποια πράγματα μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες και τι είναι εκτός των ομοδιοτήτων μα. Äh, Ευχαριστώ πολύ, Αν. Ε, ήταν ευρεία η γκάμα και πολύ επικριτικά αυτά που μας είπες. Καλό που έχουμε χρόνο. Ελπίζω να μπορέσουν να απαντηθούν αυτά. Η πρώτη απάντηση θα δώσει σίγουρα η γραμματεία μας. Πάνω, τι γίνεται με τις αρμοδιότητες και θα πρέπει να συσταθεί καμιά ομάδα εργασίας, παρακαλώ. Thank τα θέματα που έθεσε η κυρία Φανλάνκερ, που είναι βάσιμα. ο πρόεδρο τη Επιτροπή ΣΥΜΚΟ, ε, μαζί με τον πρόεδρο τη δική μα Επιτροπή, ζήτησε τη δημιουργία μια ε, ομάδα εργασία που δεν δέχτηκε η ΕΝΔΗ που ήθελε μια πιο χαλαρή μορφή συνεργασία μεταξύ του εισηγητή και των ε, σκιωδών εισηγητών και επομένω δεν έχουμε... Και επομένως δεν έχουμε συμφωνία για τα άρθρα ή τμήματα των άρθρων που να τα δέχονται οι επιτροπές. Υπάρχει όμως η έγκριση που δίνεται από τη διάσκεψη των Προέδρων για την ενισχυμένη συνεργασία βάσει των τομέων που εντοπίσαμε, ε, που εντόπισε μάλλον το αίτημα του Προέδρου. Όταν ψηφίσουμε στην Επιτροπή, ο Πρόεδρος θα στείλει μια επιστολή στον Πρόεδρο της ΕΜΒΗ και θα του ζητήσει να μην ψηφίσει για τις συγκεκριμένες τροπολογίες που εμπίπτουν σε αυτούς τους τομείς και να ψηφίσει για τις υπόλοιπες τροπολογίες. Ε, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και τροπολογίες που να εμπνέουν είναι πολύ σημαντικές. Μάλιστα, αυτή ήταν η ερώτηση προς τη γραμματεία. Η κυρία Τοματσεύσκα τώρα για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ στους μηχανισμούς αποζημίωσης. Και κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει είναι η δυνατότητα που έχει κανείς να ε, νοσηλεύεται στο εξωτερικό. Και μιλώ για τις τροπολογίες 43, 52, 104 συγκεκριμένα και όλες εκείνες που αναφέρονται σε αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα είναι τι είδους περίθαλψη θα είναι αυτή, ε? θα είναι η ίδια θεραπεία ακριβώς ή που θα έχει ταυτόσημα ή τα ίδια αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι τροπολογίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την Πολωνία. Επειδή δεν είμαι γιατρός, δεν θυμάμαι ακριβώς για ποια ασθένεια επρόκειτο. Ήταν ένα παιδιατρικό νόσημα ένα πρόβλημα που έχουν τα παιδιά ε, όπου είναι πολύ σκληροί οι μυς τους, ε, ένας δεν ξέρω ίσως είναι σπαστικό νόσημα και δεν μπορούν να περπατήσουν σωστά. Στη Γερμανία γίνονται και εγχειρήσεις και θεραπείες υπάρχουν και ε, αντιμετωπίζεται η ασθένεια αυτή. Από ό,τι φαίνεται και στην Πολωνία υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα Και γι' αυτό οι Πολωνοί δεν δίνουν ε, έγκριση ε, για αποζημίωση των ε, εξόδων νοσηλείας και θεραπείας και εγχείρηση στη Γερμανία. Αλλά στη Γερμανία δεν κάνουν μόνο την εγχείρηση, ακολουθεί και φυσιοθεραπεία, παρακολούθηση μέχρι την αποκατάσταση, την πλήρη του ασθενούς. Και έτσι το παιδί πραγματικά παραμένει μετά την εγχείρηση ε, σε περίθαλψη, παρακολούθηση και θεραπεία για να μπορέσει στη συνέχεια να ενταχθεί στην κοινωνία κανονικά. Στην Πολωνία αυτή η συνέχεια δεν δίδεται. Και υπήρξε ένα περιστατικό, ε, μια ε, κοριτσάκι 8 χρονών χειρουργήθηκε αλλά η χείριση απέτυχε. Και τώρα είναι ήδη πολύ αργά και έχασε την ευκαιρία για να περπατήσει αυτό το παιδί να λειτουργεί κανονικά στη ζωή του. Γιατί δεν του δόθηκε η απαραίτητη προσοχή μετά την εγχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι όταν μιλάμε για ορισμού και κάνουμε διατυπώσει τέτοιε στι τροπολογίε. Αυτή η οδηγία θα μπορούσε να λύσει τέτοιου είδου προβλήματα. Ελπίζω να μας οθήσει σε μια σωστή απόφαση μετά από σκέψη αυτή η οδηγία. Και όταν μιλάμε για αποζημίωση και των ιατρικών εξόδων που είναι υποχρεωμένος κανείς να καταβάλει σε μια τρίτη χώρα ή σε μια χώρα μέλος, συγγνώμη. Κάτι άλλο σημαντικό είναι στην κυκλοφορία των ασθενών να έχουμε υπόψη μας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στα διάφορα κράτη-μέλη. Να έχουν βέβαια για γιατροί πρόσβαση αλλά νομίζω αυτό ξεφεύγει από το θέμα μας. Είναι πιο ευρύτερο ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πολλές ερωτήσεις. Ο εισηγητής μας έχει το λόγο. Ο κύριος Μπραγκέτο δεν ζήτησε κανένας άλλος, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, ήλες. Α, η κυρία Σίνοτ. κυρία Σίνοτ. Πάνω στο νήμα και βέβαια έχετε το λόγο. Έχω ζητήσει το λόγο εδώ και ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ε, μερικά σχόλια ε, για τις τροπολογίες. Ανησυχώ λίγο για την τροπολογία 46. Γενικά ανησυχώ και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την προέγκριση που έτσι παρισφρεί ξανά στο σύστημα. Γιατί στη χώρα μου μας λένε ότι έχουμε το δικαίωμα να πάμε σε άλλη χώρα για περίθαλψη εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην Ιρλανδία. Ακριβώς όμως λόγω της προέγκρισης, ακόμα και αν δεν υπάρχει ε, η θεραπεία στην Ιρλανδία, δεν μας δίνουν τη θεώρηση, δεν υπογράφουν αυτό το χαρτί και δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είμαι η εισηγητρία περιβάλλοντος και δημοσίας υγείας. Σε πολλές περιπτώσεις, λοιπόν, έτσι επισέρχεται υπογείως η προέγκριση και στο άρθρο 47 μπορούν οι αρχές, ακόμα και οι τοπικές ή οι κρατικές, να ορίσουν αν υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας. Μα ακριβώ αυτό ισχύει και τώρα και δεν αφήνουν τους ασθενείς να κυκλοφορούν και μετά να αποζημιώνονται, όπως κανονικά θα ε, δικαιούνται στην ίδια τους τη χώρα. Αν θέλετε να υπάρξει αυτή η δυνατότητα, να μπορούν να πηγαίνουν στο εξωτερικό για τη θεραπεία τους οι ασθενείς, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με οποιαδήποτε μορφή πρώτερης έγκρισης από τις τοπικές μάλιστα αρχές. Γιατί στην Ιρλανδία έχουμε πάρα πολύ ε, δύσκολη εμπειρία, είναι πολύ δύσκολο να εγκριθεί καν αυτή η ε, δυνατότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρακέτ, έχει το λόγο για να ολοκληρώσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συνοδέλφους ε, που συνεισέφεραν. Ε, μου επιτρέπουν αυτά τα σχόλιά τους να προβώ σε περαιτέρω διευκρινήσεις και βελτιώσεις του κειμένου και τελικά της οδηγίας. Από τις συζητήσεις ε, που έχουν γίνει, από τις επαφές που είχα αυτή την περίοδο, πιστεύω ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της πρώτης εφαρμογής. Θα χρειαστεί μάλλον χρόνος και χρόνος για να γίνει και μία αναθεώρηση των μέσων ε, με τα οποία θα εξασφαλίσουμε αυτό το δικαίωμα που αναφέρει η οδηγία. Πάντως νομίζω ότι οι περισσότερες ε, τροπολογίες της κυρίας Λίν ως προς την γενική τους ιδέα έχουν γίνει δεκτές. Όπως και ένα τμήμα των ισχυών Βαν Λάγκε επίσης νομίζω διασκεδάζονται, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο το θέμα των μηχανισμών αντιστάθμισης, καθώς και της ε, πρώτερης ε, έγκρισης. Γιατί υπάρχει μία ταλάντευση ε, ανάμεσα σε αυτούς που τη θέλουν και σε αυτούς που δεν τη θέλουν. Νομίζω ότι η πρόταση της ε, Κομισιόν αλλά και του κυρίου Μπόουις με τον οποίο τα είπαμε λιγάκι είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε μια, ε, ένα σημείο ισορροπίας να αποφύγουμε τα δύο άκρια υπερβολική ελευθερία και υπερβολική, από τη μία και από την άλλη υπερβολικό περιορισμό, ας πούμε, να σταματήσουμε πάλι να δούμε μέσα σε αυτές τις δύο ακραίες θέσεις. Υπάρχει δυνατότητα να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας και συμφωνίας τελικά. Από αύριο θα ξεκινήσει αυτή η άτυπη διαπραγμάτευση ε, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτά τα πιο ευαίσθητα σημεία. Θα έχουμε μια άμεση και άτυπη, όπως σας είπα, επαφή γι' αυτό. Και θα τα ξαναπούμε έτσι άτυπα πάλι με τον κύριο Μπόουις. Γιατί πρόκειται για θέματα που πρέπει κάπου να καταλήξουμε, κάπου να συμφωνήσουμε. Ε, εμείς και η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή αποκλεί... δεν γίνεται να έχουμε τελείως διαφορετική άποψη εμείς. Γιατί πρόκειται για μια οδηγία που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών, αφορά όλους τους ασθενείς και δεν νομίζω ότι αυτές τις τροπολογίες αμφισβητούν αυτή την πτυχή. Εν θα τα θα προσπαθήσουμε να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα σημεία όλοι μαζί τις επόμενες μέρες. Όλοι οι αρμόδιοι. Ευχαριστώ. Ωραία, χρησιμοποιούμε καλά το χρόνο μας για τις συζητήσεις. Θα συναντηθούμε με την Άννη, είμαι σίγουρος. Αυτά τα σημαντικά ζητήματα θα εγκριθούν στις 11 Φεβρουαρίου και θα πρέπει να βιαστούμε λίγο και κατά τα άλλα στην Ολομέλεια λέει θα πάει τον Απρίλιο που θα είμαστε όλοι στον προεκλογικό αγώνα, οι παραμονέ τελευταίο σημείο. Μετά το 4 υπάρχει το 5 που μου είπαν ότι ακυρώθηκε, οπότε να περάσουμε στο 6. Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας είναι έκθεση πρωτοβουλίας. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ελισαπέτη Μωρά και έχει αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι έκθεση πρωτοβουλίας όπως είπατε και ο δυο, αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι το ζητούμενο είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, της κρίσης που μας πλήττει άμεσα και σφοδρά και όχι μόνο την οικονομία αλλά και τους εργαζομένους. Και η Επιτροπή μας ε, βεβαίως κατά κύριο λόγο θίγεται γιατί είναι στην καρδιά της ανασχόλησής μας οι εργαζόμενοι και τα προβλήματά τους. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στις τρεις μεγάλες κύριες ενότητες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης Οικονομίας. Έχουμε από τη μια ε, τους εργαζομένους, δηλαδή το ανθρώπινο στοιχείο, Κάντε λίγο ησυχία, ιδιαίτερα όσοι εξέρχεστε τις εκδόσεις, για να ακούσουμε την Ελίζα Μπέτ. Παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε το ευρωπαϊκό αυτό σχέδιο που έχει τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες. Πρώτο είναι οι εργαζόμενοι. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι τα εργατικά χέρια, το, το έμψυχο υλικό αυτό καθ' αυτό. Το δεύτερο αφορά τη ε, χρηματοοικονομική και διοικητική βελτίωση της λειτουργίας δηλαδή των διαφόρων ευρωπαϊκών συστημάτων για να εξασφαλίσουμε την ανάκαμψη. Και το τρίτο μεγάλο κεφάλαιο του σχεδίου αυτού είναι αυτό που στοχεύει σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της ε, οικονομίας που ε, θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη. Αυτά είναι τα τρία πεδία λοιπόν και καλύπτουν ε, δέκα περίπου ισχυρούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι ενίσχυση της απασχόλησης. Αυτό αφορά κυρίως ανθρώπους που έχουν χαμηλή ειδίκευση και είναι και πιο ευάλωτοι. Και θα πρέπει πραγματικά να προσιλωθούμε σε αυτό το στόχο. Διότι αυτοί είναι εκείνοι που κινδυνεύουν περισσότερο να πληγούν από την κρίση. θα κάνουμε σημαντικές επενδύσεις και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρώπη συνολικά, αλλά η πρώτη επένδυση είναι η επένδυση στο έμψυχο υλικό, στους ανθρώπους και η αύξηση των προσόντων και των ε, δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων. Γι' αυτό υπάρχει το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που γνωρίζετε ότι ε, θεσπίστηκε μετά από πρόταση της Ροζελίν Μπασλό και μπορούμε να αλλάξουμε τον προσανατολισμό του, να, να υπάρξει κάποια ανακατάταξη εκεί των κονδυλίων ε, προς την κατάρτιση των εργαζομένων. Πάντα στον ίδιο στόχο, υποστήριξη δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού μας, αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο φιλοδοξεί να μειώσει τις κοινωνικές εισφορές ε, των χαμηλομίσθων. Και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από εκεί θα δοθούν στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση των εργαζομένων. Δεύτερο μεγάλο πεδίο δράσης, είπαμε, είναι η βελτίωση της λειτουργίας και της διοίκησης και τα χρηματοοικονομικά δηλαδή πιο εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση ειδικά των επιχειρήσεων ε, μετά από χρηματοδότηση με δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από την άλλη με ενίσχυση όχι των μικρών αλλά των μεσαίων επιχειρήσεων πάλι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 30 δις είναι το πρώτο κεφάλαιο και ένα δις το δεύτερο. Και γενικά υπάρχει η βούληση απλούστευσης, απλοποίησης των διαδικασιών για να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις ενισχύσεις και στη χρηματοδότηση εταιρείε. Πάντα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θέλουμε να μειώσουμε το διοικητικό κόστος και τη γραφειοκρατία. Ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο να μπορεί κανείς να ανοίγει μια εταιρεία μέσα σε τρεις μέρες. Όλοι μας το επιθυμούμε και τον ηρευόμαστε. Είναι στόχος ε, πολύ φιλόδοξος και μεγαλόπνος και υπάρχουν και μέσα που διευκολύνουν τη ζωή των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και επίσης να υπάρχει δυνατότητα ίδρυσης εταιριών με ίδια κεφάλαιο ενό ευρώ. Τώρα, ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι κλάδοι και έρχομαι στο τρίτο που ενισχύονται και προσέχονται ιδιαίτερα. Πρώτος μεγάλος ε, κλάδος που θα πρέπει να προσέξουμε είναι με πολύ γενναίες επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών μας υποδομών. Και εδώ μιλώ και για τις μεταφορές, αλλά και για τις νέες τεχνολογίες. Και εκεί ε, υπάρχουν βέβαια τα μεγάλα έργα, τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Γιατί αν, μιλάμε για σχέδια από την αρχή, για έργα από την αρχή, από το μηδέν, ε, θα προχωρήσει η κρίση και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ανάκαμψη. Λοιπόν, θέλουμε να επιταχύνουμε τη χρήση ε, των ε, διαρθρωτικών ταμείων κυρίως του κοινωνικού ταμείου. Δηλαδή, επιτάχυση των μεγάλων έργων και των υποδομών, νέα μεγάλα έργα για να τονώσουμε την οικονομία. Δεύτερος τομέας που θα ενισχύσει και την οικονομία και την έρευνα και την καινοτομία σήμερα είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών δηλαδή τα κτίρια να εξοικονομούν ενέργεια. Ο κλάδος της οικοδομής έχει γονατίσει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τώρα να του δώσουμε μια νέα πνοή, αλλά σεβόμενοι το περιβάλλον, εξοικονομώντας ενέργεια. Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν για να βελτιωθεί ε, το επόμενο διάστημα και τα επόμενα έτη η κατάσταση των υποδομών, του κατασκευαστικού τομέα. Τρίτος και μεγάλος κλάδος που θα πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή μας και να είμαστε άκαμπτοι είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Βέβαια μιλάω και για τη θεμελιώδη έρευνα. Και σήμερα η θεμελιώδη έρευνα θα πρέπει να είναι συντονισμένη σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα, σε μεγάλους ευρωπαϊκούς στόχους. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι πρέπει να υποστηρίζουμε και μεγάλες επενδύσεις στην εφαρμοσμένη έρευνα. Που βράχει πρόθεσμα θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε νέα προϊόντα και σε νέες εξελίξεις. Ναι, λοιπόν, στην καινοτομία, στη δημιουργία και στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων. Τα επόμενα χρόνια και μετά από αυτή την τόσο σφορδρή κρίση θα κριθούμε από τη δυνατότητα της καινοτομίας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε μια θέση ε, ελπιδοφόρα για το μέλλον στην παγκόσμια οικονομία. Υπάρχουν και δύο ακόμη τομεί που δεν επιτρέπεται να ξεχάσω, που είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, που επίσης χρειάζεται στήριξη ε, σημαντική, αλλά πάλι προς νέες κατευθύνσεις, νέες εφαρμογές Και ε, οι προσδοκίες όλες αυτές και οι φιλοδοξίες δεν αντιστοιχούν απαραίτητο με τα προϊόντα που έχουμε σήμερα στην κυκλοφορία. Ε, και εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να κάνει διαφοροποίηση στα καύσιμα που χρησιμοποιεί και ε, για άλλα στοιχεία για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. Και εκεί προβλέπονται οικονομικά εργαλεία υποστήριξης. Και τελευταίος κλάδος είναι το διαδίκτυο. Και εκεί χρειάζονται υποδομές, ευρυζωνικότητα, με πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, έτσι ώστε το σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, να, ε, να υποφελούνται και οι δραστηριότητες και οι ερευνητικές δραστηριότητες να μπορούν εκεί να αναπτυχθούν. Μέσα από όλα αυτά λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καλές είναι οι επενδύσεις στοχευμένες, αλλά πρέπει να επενδύσουμε και να στηρίξουμε το ανθρώπινο δυναμικό με αύξηση των γνώσεων, με ανάπτυξη της έρευνας, με αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης και όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα γιατί πιέζουν οι χρόνοι. Ίσως ε, από εκεί να απορρέει και η δυσκολία αυτού του σχεδίου. Όταν αρχίζουμε να συζητάμε για κατάρτιση και επανακατάρτιση των εργαζομένων, αύξηση των προσόντων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων, νέες επαγγελματικές πρακτικές, πάντα υπάρχουν κάποιοι χρόνοι ε, καθυστέρησης, αδράνειας που δεν ε, ε, συνάδουν, δεν αντιστοιχούν με τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Αυτά σε γενικές γραμμές. Και εκεί έχουμε και ένα πεδίο που μπορούμε να δράσουμε ως Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ιζαμπέτ. Ποιος? Ο κύριος Δέροσα. Ο κύριος Δέροσα. τώρα. Yeah, thank you very much. Uh, I didn't expect to be the... Α, δεν είχα καταλάβει ότι θα ήμουν ο πρώτος ομιλητής. Τέλος πάντων. Παρότι είναι μια γνωμοδότηση αυτή, είναι μία από τις πιο σημαντικές ε, γνωμοδοτήσεις ε, που έχει κάνει η Επιτροπή μας τα τελευταία χρόνια, πέντε χρόνια. Είμαστε σε μια ανεπροηγουμένου κατάσταση, παρότι η βασική έκθεση και η γνωμοδότηση θα ξεπεραστούν ε, μέσα σε λίγους ε, μήνες για το, σε σχέση με το πώς δηλαδή θα ξεπεράσουμε την κρίση. Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα αισιόδοξο, ελπιδοφόρο ότι τα καταφέρνουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες σιγά σιγά να ανακάμψουν. Και ένα πράγμα που θα πρέπει να τονίσουμε στην γνωμοδότησή μας, στην Επιτροπή Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι όχι μόνο να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, αλλά ε, να τις κρατάνε οι εργαζόμενοι αυτές τις θέσεις. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη όντως, αλλά και ο κόσμος πρέπει να μπορεί να κρατήσει ε, την αγοραστική του δύναμη. Αν χάσουν οι άνθρωποι την απασχόληση τους αν του, βρεθούν άνεργοι, ε, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο για τις ε, κυβερνήσεις των κρατών μελών. Θα πρέπει να κρατήσουμε τα λεφτά στις τσέπες των ανθρώπων, ε, να υπάρχει αίσθηση της ασφάλειας. Θα πρέπει να τονίσουμε την ε, ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία με ασφάλεια. Συγγνώμη, δεν είναι σωστό μήνυμα αυτό για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η flexicurity. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι αυτή η flexicurity, η ευελιξία με ασφάλεια σημαίνει στην πραγματικότητα έλλειψη ασφάλειας. Ε, πολλοί κόσμος δεν ξέρει αν αύριο θα κρατήσει, θα έχει τη δουλειά του, αν θα μπορεί να πληρώνει το ενυπόθηκο δάνειο, αν θα έχει σύνταξη. Επομένως, να προχωρήσουμε προς την α, άγουσα της flexicurity είναι πραγματικά λάθος πολιτική απόφαση. Θα πρέπει να ε, επενδύσουμε σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία, να πείσουμε τους κοινωνικούς εταίρους ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια αλλαγή. Στην γνωμοδότησή μας θα πρέπει να δώσουμε ε, έμφαση στην ανάγκη να κρατάμε το εισόδημά μας. Να, ενθαρρύνουμε, να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να ξοδεύουν τα χρήματα που έχουν. Και εμείς να δείξουμε ότι συντοποιούμε ότι οι συντάξεις τους ε, είναι σε δινή θέση χιλιάδες, δεν πω εκατομμύρια άνθρωποι ε, είναι ήδη σήμερα σε μια άσχημη κατάσταση, μειώνονται οι συντάξει τους και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα πολύ πιο έντονα από ό,τι κάνουμε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Η κυρία Σένετ, παρακαλώ. Υπενθυμίζω, λέει η κυρία Σίνωτ, πως ε, είμαστε Επιτροπή Απασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων. Δύο πραγματάκια. Συμφωνώ με τον εισηγητή πως ε, βάρος πρέπει να δώσουμε στην διατήρηση των θέσεων εργασίας αλλά και στα νέα μοντέλα δημιουργίας θέσεων εργασίας και μια εκστρατεία που κάνω εγώ είναι όταν υπάρχουν ε, απολύσεις υπάρχουν και αποζημιώσεις και οπωσδήποτε μια κυβέρνηση που δεν έχει έσοδα το βλέπει αυτό ως πηγή εσόδων φόρου εισοδήματος. Πρέπει δηλαδή να αφήσουμε τους ανθρώπους να βοηθηθούν. Και εκεί όπου λαμβάνουν αποζημίωση οι άνθρωποι ή κάποια πρόορη συνταξιοδότηση να τους επιτρέψουμε να τη χρησιμοποιήσουν είτε για να επανεκπαιδευτούν ή για να κάνουν κάτι για να βρουν μια άλλη δουλειά και αν μπορούν να το αποδείξουν αυτό ας κρατήσουν αυτά τα λεφτά δεν είναι ανάγκη να τους τα παίρνουμε κιόλα, γιατί είναι ίσως η μόνη ευκαιρία που έχουν να μπορέσουν να βρουν μια άλλη δουλειά και αν ξέρουν ε, πως ε, θα λάβουν είτε ε, αποζημίωση για την απόλυση ή κάτι άλλο και ξέρουν ότι αυτά θα πάνε είτε στην εφορία είτε για μια άλλη δουλειά, θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργητικότητά τους για να κάνουν ε, κάποια μικρή επιχείρηση, να συνεταιριστούν με άλλους ε, πρώην συναδέλφους τους και να ανοίξουν μια άλλη επιχείρηση. Οπότε μπορούμε να ενισχύσουμε τις νέες επιχειρήσεις με το να αφήσουμε τους ανθρώπους ε, ήσυχους να βοηθούν. Και σε άλλες χώρες όπως και στη δική μου που υπάρχουν δημοσιονομικά προβλήματα οι πιο ευπαθείς ε, πάντα χάνουν τις υπηρεσίες που τους παρέχονται αλλά τα έχω πει είτε μιλάμε για τους ηλικιωμένου είτε για τους ανάπηρους οι υπηρεσίες αυτές είναι υπηρεσίες έντασης εργασίας και αν είναι να παραμείνουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους, να έχουν την αγοραστική τους δύναμη για να κινείται η οικονομία. Το να κόψουμε τις υπηρεσίες έντασης εργασίας είναι άσχημη ιδέα. Και για κοινωνικούς λόγους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι ευπαθείς και χρειάζονται τις υπηρεσίες, αλλά και επειδή μειώνεται η απασχόληση. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε εδώ πέρα... Ε, με τους εξή όρους, να, περιφρονούν, να περιφρονούνται, με συγχωρείτε, αυτά τα κονδύλια που πηγαίνουν τουλάχιστον στις πιο ευπαθείς ε, ομάδες. ευχαριστώ. Η κυρία Τόμασεύσκα έχει τον λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ενίσχυση των εργαζομένων, πάντα. Αλλά η αμοιβή των εργαζομένων ε, συνδέεται με τη ζήτηση ε, στην ελεύθερη οικονομία. Ε, αλλά το θέμα είναι ότι η οικονομία τονώνεται και από την κατανάλωση και όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα στις τσέπες τους να δαπανίσουν η ε, οικονομία αποτελματώνεται. Και θα πρέπει να τα λέει και η έκθεση αυτά. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην κατάσταση στα πολωνικά ναυπηγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει τα ναυπηγεία αυτά και να απολύσει τους εργαζομένους. Και πάμε και αγοράζουμε από τις χώρες της Ασίας ε, πλοία. Ενώ οι Πολωνοί εργάτες των ναυπηγείων λαμβάνουν αποζημίωση και επίδομα ανεργίας. Δηλαδή τους πληρώνουμε για να μην κάθονται, να μην κάνουν τίποτα, να παραμένουν σε οικονομική αδράνεια και απραξία και, να είναι εκτός οικονομίας. Όταν παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να έχουμε πάντα επίγνωση των συνεπειών. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση αυτή, ιδιαίτερα όταν σοβεί αυτή η τεράστια οικονομική κρίση παγκοσμίω. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια σφάλματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. <clears throat> Äh, Ευχαριστώ. Εγώ έχω ένα ερώτημα προς την εισηγήτρια. Εμείς στη Γερμανία έχουμε αυτές τις λεγόμενες ζώνες ε, προστασίας. Μία είναι για τις τράπεζες, μία είναι στην πραγματική ε, οικονομία. Πολλοί θεωρούν πως βεβαίως δεν υπάρχει ζώνη προστασίας για τους πολίτες για να μπορούν να εργαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να υπάρχουν και θέσεις εργασίας και ένα μέτρο είναι να φροντίσουμε από το επίπεδο του κράτους να μπορεί να βρεθεί κάποια βραχυπρόθεσμη εργασία, να παρεμβεί το κράτος και μετά να υπάρχουν ε, εργαζόμενοι οι οποίοι θα έχουν εκπαιδευτεί στην πιο σύγχρονη στο πιο σύγχρονο επίπεδο της τεχνολογίας, γιατί υπάρχει και αυτό το τεράστιο κενό για τους εξειδικευμένους εργαζόμενους. Και δεύτερο, βεβαίως, νομίζω υπήρχε και αυτή η πρόταση της γαλλικής ε, Προεδρίας Συμβουλίου που είπε ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή οικονομική κυβέρνηση Βεβαίως αυτό ήταν αντικείμενο κριτικής ε, και στη Γερμανία γιατί λένε πως είναι πολύ διαφορετικές ε, πραγματικότητες αλλά νομίζω μπορούμε να το πούμε αυτό και σε ευρωεκλογέ, ότι το αντιμετωπίσαμε αυτό από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούμε τελικά χρειαζόμαστε μια τέτοια Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση είχε δίκιο η Άγγελα Μέρκελ όταν είχε πει όχι και τελικά υπήρξε μια συνεννόηση. Νομίζω ήταν καλή αυτή, αυτός ο δρόμος που ακολουθήθηκε. Νομίζω πως η Κομισιόν το παρεκπροσωπείται επίση με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει το λόγο. Thank you very much, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστούμε και την εισηγήτρια. Σαφώς είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση, υποφέρει η ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό επηρεάζει πολλούς τομείς, αναφέρεται και αυτοκινητοβιομηχανία, η οικοδομή κτλ. Είναι πολύ χαμηλά η εμπιστοσύνη στην αγορά και η ανάλυση μας δείχνει πως θα, επηρεαστούν και, θα επηρεαστεί και η αγορά εργασίας. Και είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την ενδιάμεση πρόβλεψη της ε, Κομισιόν. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι πως ε, το ότι παίζει συνεχώς, το ότι παίζει συνεχώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ε, συνδέεται βεβαίως και με την πτώση στην αγορά εργασίας φέτος και του χρόνου. Οπότε οι προτάσεις αυτές που έγιναν και συζητήθηκαν στην Επιτροπή σας για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα της ε, κοινωνικής ένταξης, ε, ενίσχυσης επιχειρήσεων, πιο γρήγορης απελευθέρωσης κονδυλίων, στοχευμένη παρέμβαση με τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά και το ζήτημα της ευελιξίας με ασφάλεια. Κατά την άποψή μας, η ευελιξία με ασφάλεια είναι μια πολιτική σωστή που πρέπει να την υπερασπιστούμε. Επίσης και άνθρωποι που έχουν μόνιμες θέσει εργασία αντιμετωπίζουν ε, τα ζητήματα αυτά της ε, αναδιάρθρωσης ε, και αυτοί χρειάζονται και τα λοιπά Όχι μόνο όσοι έχουν τις λεγόμενες μη τυπικέ θέσει εργασία. Το βασικό είναι να συνεχίσουν να εργάζονται οι άνθρωποι. Μείωση του χρόνου εργασίας λοιπά, Είναι σαφώ απαραίτητα μέτρα Και πρέπει να κοιτάμε επίσης τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη, το τι αναφέρεται στο σχέδιο ανάκαμψης, το τι κάνουν αυτά τα μέτρα για την ε, ε, ζήτηση και μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις αλλά να δούμε και το τι γίνεται στον τομέα του προϋπολογισμού δηλαδή να έχουμε μέτρα τα οποία δουλεύουν και είναι και οικονομικά Θεωρούμε λοιπόν πως με τις προτάσεις αυτές που γίνονται, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις προτάσεις Κομισιόν, το Κοινοβούλιο κάνει ένα βήμα προς τα μπρος. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπερνάρ ντε. Είναι δυνατόν να ξεχάσουμε μεγάλο, να παραβλέψαμε μεγάλο συνάδελφο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Νόμιζα ότι με είχατε δει. Εν πάση περιπτώσει. Ε, σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μωρά για την ποιότητα της έκθεσης της και τη παρουσίασή της. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω το εξή: Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι ε, πάρα πολύ κρίσιμη. Ιδιαίτερα κρίσιμη. Κατά τη διάρκεια του έτους και ακόμα χειρότερα του χρόνου στις χώρες μας και πάλι θα φτάσουμε σε επίπεδα ανεργίας που εδώ και χρόνια μερικοί είχαμε εγκαταλείψει. Και αν σήμερα δεν το αντιληφθούμε αυτό και δεν κάνουμε κάτι, δεν λάβουμε τα χέρια τα μέτρα, τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τώρα συζητάμε τι χρώμα θα έχουν τα σωσίβια ενώ βουλιάζουμε. Είναι επίγουσα η κατάσταση. Κοιτάξτε, το συζητήσαμε πριν από λίγες μέρες στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Είναι πολύ σημαντική η κατάρτιση, η μετεκπαίδευση, η επανακατάρτιση για ε, νέες ανάγκες θα χρειαστούν πάρα πολλές προσπάθειες στην κατάρτιση των εργαζομένων και ήδη από τώρα θα πρέπει να δράσουμε. Το δεύτερο στοιχείο, η ευελιξία με ασφάλεια, flexicurity. Εγώ τίνω να πιστεύω ότι σήμερα αυτοί που μιλάνε για τη flexicurity είναι αυτοί που έχουν εγγυημένες θέσεις μόνιμες, δηλαδή δημόσιοι υπάλληλοι οι μισθωτοί ανησυχούν σε όλες τις χώρες. Και καλό θα ήταν να μην πολύ χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις, αν δεν θέλουμε πραγματικά να πανικοβάλουμε μαζικά τον κόσμο. Τρίτο, ε, με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό που είπε για τις μικρομεσαίες η κυρία Μόρα. Εκεί πραγματικά έχουμε κοιτάσματα ουσιαστικά δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Και μόνο προτείνοντας ε, συστήματα ενίσχυσης της μικρομεσαίας θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Ας πούμε δύο θέσεις απασχόλησης κάθε μικρομεσαία επιχείρηση χωρίς εργοδοτικές εισφορές. για ένα αλφα διάστημα και μέχρι να αρχίσουν να αποδίδουν αυτές οι θέσεις απασχόλησης στο εσωτερικό της ε, επιχείρησης να μην υπάρχουν εργοδοτικές εισφορές. Θα προτείνω λοιπόν εγώ μέσω τροπολογίες οι χώρες της Ευρωζώνης να προσφύγουν σε δάνειο από κοινού όμως όλες ε, με αλληλεγγύη και από εκεί και πέρα κάθε χώρα βλέπει πώς θα χειριστεί το μερίδιό της. Γιατί το ζητάω αυτό. Γιατί είδαμε ότι μερικές χώρες ε, έχουν δει ε, την πιστοληπτική τους ικανότητα να υποβαθμίζεται από τους οργανισμούς βαθμονόμησης. Οι χώρες που είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση θα έχουν και μεγαλύτερη δυσκολία να ε, δανειστούν χρήματα και τα επιτόκια θα είναι όλο και πιο υψηλά. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν αλληλεγγύη ευρωπαϊκή από την Ευρωζώνη με ευρωπαϊκό δάνειο εγγυημένο για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο στην τόσο κρίσιμη κατάσταση που έχουμε περιέλθει. Ευχαριστώ. Η συγκήτριά μας. Παρακαλώ. Ελίζαμπετ Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τα σχόλια από τους συναδέλφους μου όλα τα σχόλια. Για να συνοψίσω τα όσα άκουσα, πολλοί από εσά τόνισαν τη σημασία της εμπιστοσύνης, την οποία θα πρέπει να προωθήσουμε στους πολίτες μας. Πολλοί από εσά ε, για αυτό το λόγο ε, επιχειρηματολόγησαν με διαφορετικά επιχειρήματα. Αυτή η εμπιστοσύνη όμως ε, περνάει κάτι που δεν είχα πει πριν, ε, και μέσα από το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Γιατί τα σχέδια όπως αυτό, με αυτή τη θέληση μετατροπής, ε, αύξησης των προσόντων, θα πρέπει να διαμορφωθεί μέσα από το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έχετε παρατηρήσει ότι εγώ η ίδια δεν χρησιμοποίησα τον όρο ευέλιξη ασφάλεια. Ευέλιξία με ασφάλεια στην ε, σύνοψη που έκανα. Καταρχήν. Ε, εσείς το κάνατε. Το λαμβάνω υπόψη μου. Νομίζω ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε άλλους τρόπους αντιμετώπισης της απασχόλησης ε, ιδίως ό,τι αφορά την καινοτομία που θα μας την εξασφαλίσουν α, ε, οι ενώσεις των ε, εργοδοτών. Ε, μιλάω για νέες μορφές απασχόλησης επίσης. Συμφωνώ με τα όσα είπατε κυρία Σίνοτ για την απασχόληση, για την δημιουργία άλλων θέσεων απασχόλησης, νέων θέσεων απασχόλησης, όταν βγούμε από αυτήν την κρίση, όταν βγούμε από, αυτό, αυτή την ε, ανεμοθύελα κρίσης, ανεργίας κτλ. που βρισκόμαστε, δεν θα έχουμε τις ίδιες θέσεις απασχόλησης, το ίδιο επίπεδο απασχόλησης στις επιχειρήσεις. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα πρέπει να ε, δράσουμε ε, στην εμπιστοσύνη, στις θέσεις απασχόλησης, στο επίπεδο της θέσης απασχόλησης και στο επίπεδο των επενδύσεων, με νέες λύσεις. Που τόνισαν οι συνάδελφοι. Κρατάω και αυτό που είπε η Κομισιόν επίσης. Ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τον κόσμο στο χώρο εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε μονίμως για να το καταφέρουμε. Θα λάβω υπόψη πάντως όλα αυτά τα σχόλια ε, στις προτάσεις επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. 10 Φεβρουαρίου έχουμε την συζήτηση των τροπολογιών και 11 του μηνός θα ψηφίσουμε. Εκτός αν δεν συμφωνεί ο... Κάνω όπως κάνει ο Γιάννα Άντερσον που του αρέσει να χτυπάει το σφυράκι του, ο Πρόεδρο τη Επιτροπής μας. Τώρα το λόγο έχει η Γαμπριέλα Κρέτσου που έχει επίσης ένα σημαντικό θέμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα αίτημα για σύμφωνη γνώμη, προκειμένου να τροποποιήσουμε τον κανονισμό 1083 για τους κανόνες χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής. Πρόκειται για μέτρα νομοθετικής τροποποίησης που εγγράφονται στα πλαίσια του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης, το οποίο μόλις τώρα συζητήσαμε. Τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν αυτή την πρόταση ομόφωνα Τώρα, σε τι συνίσταται αυτή η πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων. Υπάρχουν επίσης ε, τροπολογίες για τις επιλέξιμες δαπάνες, για τα ανώτατα όρια για τις προκαταβολές μπορούν να κάνουν εκείνοι που δίνουν αυτά τα ταμεία, τα, τις δόσεις προχρηματοδότησης τις οποίες αυξήσαμε, σε διαφορετικό ποσοστό στα παλιά κράτη-μέλη και σε διαφορετικό ποσοστό στα καινούργια κράτη-μέλη. Συνολικά πρόκειται για μια απλούστευση επίσης των διαδικασιών. Η οικονομική επίπτωση φτάνει στα 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα θέλαμε να δεχτείτε τη σύμφωνη γνώμη με κάποιες επιφυλάξεις, να γίνει δεκτή μάλλον η σύμφωνη γνώμη. Δεν μπορούμε αυτές τις επιφυλάξεις να τις συμπεριλάβουμε εδώ, γιατί πρόκειται για σύμφωνη γνώμη, αλλά θα ήθελα να τις αναφέρω παρόλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό τα κονδύλια να ξεμπλοκάρονται πολύ πιο γρήγορα. Επίσης θα πρέπει οι στόχοι να υλοποιηθούν. Έχουμε υπόψη μας την κοινωνική συνοχή, την διευκόλυνση πρόσβασης στην ομάδα εργασίας. Θα είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον, δεδομένων όλων αυτών των μηνυμάτων κρίσης, το να υποστηρίξουμε επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το να χρησιμοποιήσουμε τους ε, τοπικούς πόρους αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική στόχη. Όμως, αυτή η, πρόταση είναι μία, θα έλεγα, επιταγή εν λευκό. Θα πούμε ναι, γιατί είναι μία πρόταση χρήσιμη για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, αλλά δεν έχουμε κανέναν έλεγχο όμως για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα ήθελα να συνάγω όμως και ένα θετικό συμπέρασμα εδώ. Υπάρχει ένα προηγούμενο το οποίο δημιουργείται έτσι και θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στο μέλλον αυτό το προηγούμενο. Πολύ συχνά στο παρελθόν οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής μας που αφορούσαν τα κοινωνικά θέματα ξεχνιούνταν γιατί δεν είχαμε κατάλληλη νομική βάση για τέτοια προγράμματα, για να τα προωθήσουμε. Μετά την έγκριση όμως αυτού εδώ του κειμένου, νομίζω ότι θα γίνει σαφές ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση θα βρίσκεται πάντα και η νομική βάση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως. Μαρία Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτοπούλου, έχει το λόγο. Τι όνομα είναι αυτό δύσκολο. Μεσή, Τόμας. Ε, ε, ε, συγχαίρω την ε, συνάδελφο Κρατσού για την ε, αποδοχή της κοινή θέση και συμφωνώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε από κοινού και με αμοιβαία εμπιστοσύνη γιατί πράγματι στον έλεγχο της διανομής δεν μπορούμε να έχουμε άμεση πληροφόρηση και πρόσβαση και να δώσουμε μια ενθάρρυνση στα κράτη-μέλη να συγχρηματοδοτούν και να χρησιμοποιούν τα ταμεία, να μην αφήνουν να χρησιμοποιείται ε, τα ποσά που τους ε, δίνονται, αλλά να τα ε, διαθέτουν ε, με τη συγχρηματοδότηση και με διαφάνεια και ε, καλή ε, διακυβέρνηση για το όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ Μαρία και συγχαρητήρια. Χτες είχατε λέει πρωτοχρονιά λέει ο πρόεδρος που μας έχει για ε, αργά βέβαια, αλλά ε, καλή χρονιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Λίγα πράγματα έχω να πω. Ε, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε αυτή την πρόταση. Είμαστε πεπισμένοι πως είναι μια σημαντική πρόταση που γρήγορα θα οδηγήσει στο να επιταχυνθούν οι δημοσιονομικές ροές στα κράτη-μέλη και άρα σε τελική ανάλυση να αυξούν οι χρηματικές ροές στους ανθρώπους που εφαρμόζουν αυτά τα έργα. Αναφέρατε κύριε εισηγήτρια πως δεν είστε τόσο ικανοποιημένοι με το ότι ε, θα γίνει αυτό χωρίς δικό σας έλεγχο. Δεν θα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα γιατί τα προγράμματα τα οποία ε, αλλάξαμε με τα κράτη-μέλη δεν αλλάζουν με αυτή την αλλαγή του κανονισμού και θα πρέπει βεβαίως να συνεχίσουν να εφαρμόζονται με πλήρη διαφάνεια και από τα κράτη-μέλη και από τις περιφέρειες και ελπίζω πως ε, με την πρόταση αυτή δεν θα χαθεί τίποτα από πλευράς κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για αυτή την έκθεση και ελπίζω πως ε, με αυτή την ε, αλλαγή θα οδηγηθούμε στην ε, αλλαγή του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα μπορέσουμε σύμφωνα να σύντομα με να συμφωνήσουμε τα τις με τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε. Μαρία, κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις έχετε να κάνετε ή τελειώσαμε. Παρακαλώ, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, λέει κυρία Κρέτσο. Σίγουρα, ως βουλευτές, εμείς εδώ εκπροσωπούμε τους πολίτες των κρατών μελών και υποστηρίζουμε βεβαίως την πρωτοβουλία αυτή, διότι πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμη για τους πολίτες. Δεν έχουμε γενική αντίρρηση και καταρχήν, αλλά για τη διαδικασία μιλώ και νομίζω ότι θα δημιουργήσει και γνωρίζουμε ότι θα δημιουργήσει προηγούμενο. Και ίσως το ξαναβρούμε μπροστά μας. Αλλά ελπίζω η στόχοι να είναι σαφείς και ελέγξιμοι. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους. Σε ευχαριστώ κυρία Κρέτσου. 29 Ιανουαρίου είναι αυτή τη βδομάδα δηλαδή η προθεσμία για τις τροπολογίες και θα το συζητήσουμε το θέμα βεβαίω 11 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ. Επόμενο σημείο, το σημείο 8, κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη. Έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών. Κυρία Μαδίρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στόχος αυτής της ε, γνωμοδότησης ε, για την ε, Επιτροπή Ελευθεριών είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό. Ήταν ήδη πολύ σημαντικό αυτό πριν πέρα ράσουμε στην οικονομική κρίση, αλλά βεβαίως το θέμα αυτό γίνεται ακόμη σημαντικότερο τώρα γιατί όλοι ξέρουμε πως η βιωσιμότητα του συστήματός μας σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την δυνατότητα απορρόφησης νέων μεταναστών. Εάν σκεφτούμε πως ε, γύρω στα 50 εκατομμύρια άνθρωποι θα καταλήψουν ε, μέχρι το 2060 τον εργαζόμενο πληθυσμό. Βλέπετε πως έχουμε μια απειλή στο σύστημα. Οπότε ήδη η μετανάστευση πρέπει να θεωρείται σημαντική πρόοδος και όθηση για την οικονομία είναι ξεκάθαρα τα συμπτώματα της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι ξεκάθαρα ζήτημα διαχείρισης ε, του, της μετανάστευσης και του δυναμικού που παρουσιάζει. Τα ζητήματα βεβαίως που προκύπτουν δεν είναι πάντα τα καλύτερα και τα ερωτήματα δεν είναι πάντα τα καλύτερα αυτά τα οποία διατυπώνονται. Όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχει σοβαρό οικονομικό δυναμικό στη μετανάστευση αλλά γνωρίζουμε πως οι δυνατότητες πρόσβασης στην εργασία, της κατάρτισης, της συνταξιοδότησης κτλ. δεν έχουν οργανηθεί με τον αντικειμενικά καλύτερο τρόπο. Επίσης γνωρίζουμε πως όλοι είμαστε κατά της παράνομης εργασίας γιατί αυτό ε, παραβιάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά επειδή αυτή γίνεται κατά κύριο λόγο προσφέρεται από τους μετανάστες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί υπάρχει και το ζήτημα της επισφαλούς ε, εργασίας ε, η οποία είναι ιδιαιτέρως βεβαίως ευάλωτη ως μέρος του παρόντος οικονομικού συστήματος κάτι πρέπει να θυμόμαστε αλλά πρέπει να θυμόμαστε επίσης πως οι οικονομίες αυτές είναι πολύ κοντά μας, ε, στη γειτονιά μας θα έλεγα και έχουν τεράστιο στο ανεργίας και έλλειψης ευκαιριών για τους νέους και τις γυναίκες. Ειδικά αν δούμε γύρω-γύρω στη Μεσόγειο, ε, όπου είναι προφανές ότι αυτό συμβαίνει. Και το ίδιο ισχύει και για την υποσαχάρη Αφρική. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε προς αυτά τα σύνορα και να κοιτάμε τη μετανάστευση όχι μόνο από πλευράς ασφάλειας, πρέπει να θυμόμαστε πως μιλάμε για ανθρώπους και πως υπάρχει εδώ πέρα αμοιβαίο όφελος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις χώρες εταίρους. Αμοιβαίο όφελος λοιπόν από τη διαδικασία αυτή της ε, μετανάστευσης. Βεβαίως σαφώς προκύπτει και το ζήτημα που δεν έχει λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το πώς θα βρούμε ποιες είναι οι δεξιότητες τους και οι άτυπες ε, και τα προσόντα τα οποία έχουν τυπικά πράγματα, τα οποία ε, δύσκολα τα έχουμε και για τους δικούς μας ε, πολίτες αλλά πρέπει να τα δούμε και για τους μετανάστες, δηλαδή το τι μαθαίνουν όταν έρχονται εδώ πέρα και το τι είχαν μάθει και στις χώρες τους πριν ξεκινήσουν, γιατί είναι δεξιότητες αυτές δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Καθώς αρκετά οι δεξιότητες χαραμίζονται όταν βλέπουμε το πού δουλεύουν οι μετανάστες. Επίσης ε, η ιδέα αυτή της διαβίου εκπαίδευσης πρέπει να είναι και δικαίωμα εγγυημένο των μεταναστών εκτός από των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό, πρόσβαση στη μάθηση της γλώσσας της χώρας όπου μένουν και επίσης να υπάρχει και μια κοινωνική ενσωμάτωση εκτός από την εργασιακή. Ε, είμαι σίγουρη πως μια τέτοια πολιτική θα επιτρέψει την εφαρμογή της ε, πολιτικής ίσων ευκαιριών και το να αποφευχθούν ε, οι διάφορες υπεκφυγές που χρησιμοποιούνται για να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή Χρειαζόμαστε ξεκάθαρες και διαφανείς διαδικασίες για να μπορούν οι μετανάστες να βρίσκουν δουλειά ανάλογη των προσόντων τους. Υπάρχει πίεση βεβαίως στα σύνορά μας και το γνωρίζουμε αυτό, κάτι το οποίο μπορεί να απογοητεύσει τους ε, ανθρώπους. Γνωρίζουμε πως ε, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ε, έρχονται εδώ πέρα και ψάχνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Χίνα που κάνει τα χρυσά αυγά. Και πολλές ευκαιρίες ε, που θα μπορούσαν να τις εκμεταλλευτούν στις δικές τους ε, χώρες που προκύπτουν από επενδύσεις μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τις ε, εκμεταλλεύονται αλλά παραμένει αυτό το κενό αν θέλετε των προσδοκιών ακόμη και μεταξύ των 27 κρατών μελών υπάρχει αυτό το λεγόμενο το, το το δίκτυο που καλό θα ήταν να επεκταθεί και σε τρίτες ε, χώρες. Ε, Δηλαδή να μπορούν τα κράτη-μέλη να αναζητούν ανθρώπους με συγκεκριμένες δεξιότητες και να μπορούν να τους αναζητήσουν σε τρίτες χώρες. Και με αυτό τον ε, τρόπο δεν θα ξεκινάνε οι άνθρωποι χωρίς να ξέρουν πού θα καταλήξουν και να περιμένουν ε, να, να βρουν δρόμους στρωμένους με χρυσάφι και να μπαίνουν ε, στις βάρκες και ό,τι γίνει θα μπορέσουμε έτσι να δείξουμε πως ε, ακόμα και αν δεν υπάρχουν ε, ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως υπάρχουν στις χώρες ε, προέλευσης. Οπότε και με τη χρήση των ειδικών κέντρων που έχουν ήδη συσταθεί σε ορισμένες χώρες και θα ξεκινήσουν σε άλλες και χρησιμοποιώντας και τις αντιπροσωπείες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα και να συμβουλεύουμε τους ε, ανθρώπους και ακόμα και για την ε, ύπαρξη μικροπιστώσεων, κάτι το οποίο θα του ενθαρρύνει στην χώρα προέλευσης. Και εκεί πέρα μπορεί να ενθαρρύνουμε τις δυνατότητες επενδύσεων ώστε να μην ε, ασχολούνται οι άνθρωποι μόνο με το πώς θα μπορέσουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο βεβαίως να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά όταν φτάνουμε σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο δεν υπάρχει ανάμειξη στη διαδικασία αυτή και οι ανάγκες ε, αυτές είναι μεγάλες. Πρέπει και λοιπόν και το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο να εμπλέκονται στη διαδικασία για τις πραγματικές ανάγκες αγοράς εργασίας και στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής, να μην ασχολούνται μόνο με την έλλειψη ε, εργατικού δυναμικού σε κάποιες χώρες, αλλά να δυσφαλίζουν πως ε, και οι μετανάστες μετά θα ενσωματώνονται σωστά. Υπάρχει βεβαίως μια λογική διαχείριση ε, πίσω από όλα αυτά, αλλά αυτό το οποίο είναι απολύτως σημαντικό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 dos países terceiros ou, no caso da comunidade escolar, em que sejam incluídos nas matérias curriculares a multiculturalidade e a descodificação das diferentes realidades culturais em presença. Esta é uma realidade que existe em alguns países. Όταν διασφαλίζεται a πολυπολιτισμικότητα των, διαφορε... διαφορετικών πραγματικοτήτων, πράγματα τα οποία γίνονται ήδη και χρήσιμο θα ήταν να γίνονται με, έτσι, με έναν πιο συντονισμένο τρόπο. Οπότε, όταν μιλάμε τώρα για μια κοινή μεταναστευτική πολιτική είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Είναι σαφές πως υπάρχουν ε, διαφορετικά ε, μέσα και δεν μπορούμε να έχουμε κοινή μεταναστευτική πολιτική αν δεν συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει να έχουμε και κοινή πολιτική ασύλου που θα βασίζεται ε, ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μανέρα. Η Μαρία, κυρία Παναγιωτοπούλου παρακαλώ. Ευχαριστώ Τόμας. Να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει μετάφραση γιατί η ελληνική μετάφραση είχε χαθεί στο τέλος. Υπάρχει. Γίνεται κανονικά η μετάφραση από τα ελληνικά. Ωραία. Ναι, ναι. Ε, ε η, η συγγήτρια ε, είπε πολύ περισσότερα στην ε, ανάλυση της από όσα γράφονται στην ε, γνωμοδότηση. Είναι μόνο μια γνωμοδότηση που κάνει η Επιτροπή μας προς την ε, Επιτροπή Ελευθεριών που παρουσιάζει την έκθεση πρωτοβουλίας για την ανακοίνωση της Επιτροπής. Όλοι είμαστε ευχαριστημένοι που επιτέλους έστω και με μια ανακοίνωση μπαίνει σε δρόμο η κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε όμως ότι εκτός από αυτή την ανακοίνωση υπάρχουν και συγκεκριμένες άλλες αποφάσεις που έχουμε πάρει και εδώ από αυτήν την Επιτροπή έχει περάσει γνωμοδότηση ε, για την ε, μπλε κάρτα και ε, ακολουθούν ίσως και άλλες προτάσεις. Ε, μάλιστα ε, πολύ σημαντική είναι η συγκεκριμένη εκείνη απόφαση για τα ε, πέντε ταμεία που συνοδεύουν την καινή μεταναστευτική ε, πολιτική και νομίζω πως πρέπει να αναφερθούμε και εμείς στη γνωμοδότησή μας για τη χρήση αυτών των χρηματοδοτικών μηχανισμών ε, που θα βοηθήσουν για να ε, είναι περισσότερες και καλύτερες οι ευκαιρίες απασχόλησης και των μεταναστών. Ε, πολύ σωστά παρουσίασε η, η της την, τις σχέσεις ε, και τη συντεταγμένη ε, μεταναστευτική πολιτική ε, που θα κάνει πιο ανθρώπινη την πολιτική αυτή από ό,τι είναι σήμερα που είναι ανοργάνωτη και κατά την περίσταση χρησιμοποιούμενη. Μιλούμε για χρησιμοποίηση των μεταναστών σήμερα όμως σε γαλλικό ε, περιοδικό πολιτικού περιεχομένου είδα ένα τίτλο, δεν διάβασα το άρθρο ότι οι πόλεις αδειάζουν από μετανάστες και τι θα γίνει που θα μας λείψουν ε, εργατικά χέρια. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται αυτή η κοινή πολιτική και η γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής μας είναι σημαντική γιατί αφορά την κύρια απασχόληση των μεταναστών, την εργασία. Ε, οι τροπολογίες ε, φαντάζομαι θα μας δώσουν την ευκαιρία να συμπληρώσουμε ε, γιατί όχι μόνο η αναγνώριση των προσόντων είναι βασική ώστε να χρησιμοποιείται σωστά το ανθρώπινο δυναμικό αλλά πρέπει να λυθούν και προβλήματα όπως τα, προβλήματα, τα ασφαλιστικά προβλήματα επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην παλιότερη μετανάστευση ε, όταν διμερείς συμφωνίες ε, μπορούσαν να λύνουν τα θέματα της ε, ασφαλιστικής κάλυψης και η Γερμανία είχε δώσει τέτοια καλά παραδείγματα όταν δέχτηκε πολλές χιλιάδες μεταναστών από τις σήμερα ευρωπαϊκές χώρες του Νότου ε, πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και τα παραδείγματα του παρελθόντος ε, για να ε, σχεδιάσουμε σωστά το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα βλέπουμε την ισχύ των γυναικών. Frau Power. Ακούσαμε την Τζαμίλα, τη Μαρία και τώρα την Ελιζαμπετή και στη συνέχεια την Καμπριέλα και τη Λύ. Εμείς <laughs> χαιρόμαστε. Η Ελιζαμπετ Μωρά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι αυτή η πολιτική μετανάστευσης και ρύθμισης της μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αποκτήσει σάρκα και οστά. Θα ήθελα να κάνω δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις μόνο που αφορούν την παράγραφο 4 και την παράγραφο 7. Θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω από την εισηγήτρια να μου πει γιατί χρησιμοποιεί την έκραση, έκφραση ε, εκμάθηση ε, καθ' τη διάρκεια του βίου και όχι κατάρτιση, διαβίου κατάρτιση. Γιατί μαθητεία και όχι κατάρτιση. Δεν θα πρέπει να δούμε την έννοια της ε, ε εκπαίδευσης με τον πιο ευρύ, δυνατή, ευρύ δυνατό τρόπο γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο τις τεχνικές καταρτήσεις, αλλά και άλλες μορφές εκπαίδευσης. Δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να σχολιάσω. Είναι σημαντικό να ζητήσουμε ένα συντονισμό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, γιατί στα πλαίσια της αποκέντρωσης, αυτά τα επίπεδα, το τοπικό και το περιφερειακό, έχουν σημαντικές ε, αρμοδιότητες ό,τι αφορά την κατάρτιση. Ο συντονισμός λοιπόν δεν πρέπει να γίνει μόνο σε, στο επίπεδο της απασχόλησης αλλά και σε, στο επίπεδο της κατάρτισης στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτές τις τροπολογίες θα ήθελα να ε, δω στο κείμενο που μας προτείνεται. Η κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ. Μία πιο γενική παρατήρηση έχω να κάνω. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δημιουργούμε τομεακές πολιτικές πάρα πολύ συνεκτικές, οι οποίες όμως δεν είναι συνεκτικές μεταξύ τους αυτές οι τομεακές πολιτικές. Παραδείγματο χάρη η πολιτική ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ του επιτρέπω στους μετανάστες την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ε, αγορά εργασίας και στις χώρες μας με, με σε πλαίσιο ισοτιμίας και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο να υποστηρίζω επιλεκτικά την άφηξή τους. Είτε με αυτόν τον τρόπο δημιουργώ ανταγωνισμό ε, μεταξύ αυτών ή μεταξύ αυτών και των Ευρωπαίων πολιτικών, πολιτών, συγγνώμη, είτε με αυτόν τον τρόπο προσελκύουμε τα μυαλά, τα κεφάλια, ας πούμε, και τους υπόλοιπους τους διώχνουμε. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν αυτή τη διάκριση. Η οικονομική κρίση, νομίζω, μας βάζει σε μια κατάσταση όπου θέλουμε να, φρενάλουμε, να φρονάρουμε λιγάκι την άφηξη των μεταναστών, γιατί και εμείς έχουμε προβλήματα απασχόλησης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολιτικές δεν θα πρέπει να είναι συντονισμένες και συνεκτικές. Ευχαριστώ. Η κυρία Λίν, τελευταία. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Εγώ συμφωνώ να υπάρξει μια κοινή μεταναστευτική πολιτική. Είναι κάτι που το ζητάμε για χρόνια μερικοί από εμά. Ξέρω ότι θα υπάρξουν αντιστάσεις και αντιδράσεις σε πολλά κράτη-μέλη λόγω της οικονομικής κρίσης. Πρέπει να ξέρουμε ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τις θέσεις απασχόλησης τους, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτρέψουμε σε ξένους να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι πρέπει να πάμε προς την ε, κατεύθυνση αυτή. Στο σημείο 2. Μιλάτε για τους ε, μετανάστες εργαζομένους. Νομίζω ότι αυτοί είναι Ευρωπαίοι πολίτες που μεταναστεύουν εσωτερικά. να συζητήσουμε, να ζητήσουμε τον όρο, να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, συγγνώμη, μετανάστες και όχι μετακινούμενοι, έτσι. Αυτό εννοούμε νομίζω. Μετανάστες, δηλαδή απ' έξω από τρίτες χώρες και όχι εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υποβάλω και κάποιες τροπολογίες για αυτό το σημείο 2, ούτως ή άλλως. Αυτό που είπατε για τη σπατάλη των προσόντων. Ναι, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα προσόντα. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, να βλέπουμε τι προσόντα έχουν οι μετανάστες από τις διάφορες χώρες. Δεν νομίζω ότι υποτιμούμε τα προβλήματα, τα προσόντα μόνο των γυναικών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν γιατροί που δεν μπορούν να συνεχίσουν ε, την επαγγελματική του σταδιοδρομία γιατί τα προσόντα τους δεν αναγνωρίζονται. Είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες. Και σε άλλα επαγγέλματα επίσης έχουμε αυτό το πρόβλημα. Επίση, συχνά ε, βλέπουμε ότι άνθρωποι με υπερβολικά πολλά προσόντα κάνουν ε, ταπεινότερε δουλειές. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό το θέμα, λοιπόν. Επίσης, δεν μίλησατε καθόλου ε, για την εμπορία ανθρώπων και τα θύματα αυτά. η Επιτροπή μας θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Καλό θα ήταν να αναφερθεί και κάτι για την έκθεση, ε, στην έκθεση αυτή, για αυτά τα θύματα από την εμπορία. Όχι μόνο για σεξουαλικούς λόγους, αλλά για οικιακή σκλαβιά. Για να δουλέψουν ε, στην, στον αγροτικό τομέα, σε διάφορους τομείς, σε διάφορους κλάδους, σε διάφορες βιομηχανίες. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα να μην βλέπουμε μόνο τους ε, λαθρομετανάστες, αλλά και αυτούς που τους έχουν ε, βάλει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη θέλησή τους, ως θύματα εμπορίας. Συμφωνώ με την έκθεσή σας, απλώς πρέπει να κάνουμε κάποια χτενίσματα, αν θέλετε, και κάποιες προσθήκες στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ, Steve Hughes. Για να σας αποδείξω ότι και τα αρσενικά μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ κανονικά θα ήθελα να βάλω πολύ περισσότερα πράγματα στην γνωμοδότηση όπως και η Τζαμίλα, αλλά έχουμε περιορισμούς. Ωστόσο, το εξή θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Να υπάρχει ένα σύστημα ελεγμένο και με σωστή παρακολούθηση της μετανάστευσης. Αυτό δεν είναι μόνο υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και υπέρ των κρατών προ ε, έλευσης. Κινδυνεύουν οι Φιλιππίνες να μείνουν από νοσηλεύτριες γιατί πάνε όλες και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Τελευταίος ήταν ο Στίβεν. Η Τζαμίλα έχει το λόγο για να συνοψίσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους πολύ σωστά και εύστοχα αυτά που μας είπατε. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να τα συμπεριλάβω στη γνωμοδότησή μου. Όταν μιλάμε για μια κοινή πολιτική ασύλου, ε, δεν ξέρω αν είναι του παρόντος, αν είναι εντός θέματος γιατί και εγώ ε, ε, ήταν μεγάλο ο πειρασμός και για μένα να μην το αναφέρω. Ήθελα πάρα πολύ να το βάλω, αλλά δεν το έθεσα. Είναι και σχέδιο γνωμοδότηση. Αν αρχίσουμε να συζητάμε για ε, ευρύτερα θέματα, δεν θα μπορέσουμε να τα συμπεριλάβουμε. Τα σχόλιά σα όμω, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Θα ήθελα να πω το εξή. Προθεσμία είναι πάρα πολύ σφιχτή. Αύριο το μεσημέρι στις 12. Αύριο το μεσημέρι στις 12 λέγει η προθεσμία διότι η αρμόδια επιτροπή ΛΥΜΠΕ Ελευθεριών ήδη στις 5 Μαρτίου θα ψηφίσει. Ελπίζω όλα αυτά να τα καταφέρετε, αλλά η επισηγήτρια ότι μπορεί να συμπεριλάβει αυτές τις απόψεις και ελπίζω να είναι καλή γνωμοδότηση τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Άλλα θέματα έχουμε, ερωτήσεις, συμπληρώσεις. Όχι. Επόμενη συνεδρία στη 10 Φεβρουαρίου, 3 με 6.30 και στις 11 Φεβρουαρίου πρωί και απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Λήξη συνεδρίασης.